Τώρα και τώρα περνάμε στις επεξηγήσεις ψήφου. Ξεκινάμε με την έκθεση Μπάστος και Δίνω τον λόγο στον κύριο Μπαλτασάρε. Κύριε Μπαλτασάρε, πού είσαστε. We wait uh, some minutes. Συνάδελφοι, αποχωρήστε γρηγορότερα, έτσι ώστε όποιος θέλει να κάνει δήλωση, επεξήγηση να μπορεί. Εν ειρήνη ή δυνατόν. Με ησυχία, παρακαλώ. Κύριε Μπαλτασάρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την έκθεση της συναδέλφου Μπάστος που υποστήριξα Δυστυχώς η μεγάλη χρηματοοικονομική κρίση που έπληξε την Ευρώπη είχε αρνητικές επιπτώσεις ως προς την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς από επιχειρήσεις και πολίτες ή από εθνικά κινήματα. Αυτό δυστυχώς ε, οδηγεί στην παραγνώριση της εξαίρετης αυτής εργασίας αρκεί να σκεφτείτε τη μεγάλη μεταρρύθμιση για τις δημόσιες προμήθειες ή για τις καθυστερήσεις πληρωμών. Θα πρέπει να ενισχυθεί η διαθεσμική συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών, γιατί σημαντικά μέτρα όπως μέτρα πρόληψης έχουν καθυστερήσει εξαιτίας των διαθεσμικών κρίσεων και εθνικών υπολογισμών. Θα πρέπει να έχουμε μία ενιαία προσέγγιση της διακυβέρνησης αυτής και την κατάλληλη νομοθεσία για την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και των δικαιωμάτων των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε κύριε Μπαλντασάρε. Ο κύριος Φιλίπ Ζουβέν. Πρόεδρε, νομίζω ότι στην πολιτική πρέπει να μιλάμε καθαρά. Η εσωτερική αγορά που έκλεισε τα 20 της χρόνια ε, προσέδωσε πολλά ευεργετήματα, αλλά σήμερα η εσωτερική αγορά έχει νόημα μόνο αν προστατεύσει την απασχόληση και τις βιομηχανίες μας και αν δεν αλλάξουμε τις πρακτικές μας, τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Μεγάλες ε, οι οικονομικές δυνάμεις, ε, το Κατάρι, η Κίνα, η Ιαπωνία θα υπερισχύσουν και θα αλλάξουν την έδρα τους ως προς τα βιομηχανικά τους προϊόντα μακριά από την Ευρώπη. Θα πρέπει να προωθήσουμε μια πραγματική προστασία της ε, ευρωπαϊκής, ευρωπαϊκής αγοράς, ενιαίας αγοράς, υπομορφή και προστατευτισμού. Ευχαριστούμε κύριε Ζουβά. Η κυρία Τζανίκη έχει το λόγο. Απούσα. Η κυρία Κωνσταντς Λεγκρίπ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως μέλος Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών έχω ενδιαφερθεί πολύ στην έκθεση, για την έκθεση Ρετσίνα Πάστος με βάση 20 θέματα που απασχολούν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και συζητήσαμε την έκθεση αυτή σε ε, συνεργασία με την συζήτηση, ε, σε συνδυασμό με τη συζήτηση που έγινε για τα 20 χρόνια της ελεύθερης αγοράς που επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, ανθρώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων η οποία πρέπει να ασκείται πλήρως στο εσωτερικό του χώρου ζωής μας, των ανταλλαγών και της ελευθερίας μας που είναι η εσωτερική αγορά. Ενδιαφέρθηκα ιδιαίτερα από το γεγονός ότι στο, από τα πρώτα θέματα που εξέφρασαν ως ανησυχία οι Ευρωπαίοι συμπολίτε μας είναι η δυσκολία αναγνώρισης των εμπορικών ε, ε, επαγγελματικών προσόντων και πρέπει να προλάβουμε την κατάσταση αυτή, να είμαστε αποτελεσματικοί. Αυτό ε, περιμένουν από εμά οι συμπολίτε μα για να δημιουργήσουμε στο άμεσο μέλλον μια διαδικασία αναγνώρισης των τίτλων, των επαγγελματικών τους προσόντων και των δυνατοτήτων τους με τρόπο απλούστερο, πιο αποτελεσματικό και όχι τόσο δαπανηρό. Ως του ΕΛΚ για το θέμα αυτό του εξυγχρονισμού της διαδικασίας αυτής. Εργάζομαι δραστήρια με τα άλλα μέλη της Επιτροπής ΥΜΚΟ για να ανταποκριθούμε σε αυτή τη σοβαρή πρόκληση της κινητικότητας. Περισσότερη κινητικότητα για περισσότερη Ευρώπη. Αυτό ζητούν οι συμπολίτες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Λεγκρίπ. Δίνω το λόγο στον κύριο Ρέστε Ρώση. Ευχαριστώ με την ενιαία αγορά που ήταν απαραίτητη για την πραγμάτωση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ευρώπη 2020 θα πρέπει παράλληλα να ε, προωθήσουμε την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και τη θέση των πολιτών. Υπάρχει μεγάλο χάσμα όμως μεταξύ προσδοκιών και πραγματικότητα το οποίο δημιουργεί μεγάλες ανησυχίες, ιδιαίτερα όσο προς το φορολογικό καθεστώς, την καταβολή του ΦΠΑ και ούτω καθεξής. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε την ανταγωνιστικότητα δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, προωθώντας έρευνα και ανάπτυξη και εδαφική ακαιρεότητα. Έτσι θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τα ποιοτικά μας προϊόντα. Θα πρέπει να εναρμονίσουμε το κόστος της ενέργειας που για πολλά κράτη-μέλη παρουσιάζει κάτι το δυσθεώρητο. Σε ευχαριστώ. Δίνω τον λόγο στον κύριο Ρέπο. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα την έκθεση. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για το ότι εδώ πέρα πραγματικά ενθαρρύνουμε τους επιχειρηματίες να στηρίξουν τους νέους οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό και ακριβώς εδώ πέρα πρέπει να δούμε τους ασθενέστερους επίσης ε, η Κομισιόν πρέπει να κάνει μια εκστρατεία διαφώτισης, ενημέρωσης και μια ε, μελέτη του αντικτύπου γιατί αλλιώς ε, θα ξοδεύουμε τα λίγα μέσα που έχουμε στην ε, διάθεσή μας. Νομίζω λοιπόν πως ε, θα πρέπει να βρούμε μέσα να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για περισσότερη κινητικότητα. Σας ευχαριστώ κύριε Ρέπο. Λόγο έχει ο κύριος Ντίβα. Κύριε Πρόεδρε, με τιμά το ότι διαλέξετε να μιλήσετε αγγλικά σήμερα, κατά το οποίο βρίσκω θαυμάσιο. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν 20 ανησυχίες ε, πάνω στις οποίες έχει εστιάσει ο νομοθέτης. Οι ανησυχίες αυτές είναι σημαντικές. Αφορούν ε, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, επαγγελματικά προσόντα, τα κράτη-μέλη να έχουν δικαιώματα κληρονομιάς, ε, συνταξιωτικά δικαιώματα. Αλλά αυτό το οποίο είναι πιο σημαντικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου αυξάνεται η ανεργία, είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας και ο κινητήρα δημιουργία θέσεων εργασίας είναι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Είναι η εμπροστοφυλακή τη δημιουργία θέσεων εργασία. και πάνω σε αυτό έχει εστιαστεί η έκθεση, γι' αυτό τη στήριξα. Αλλά 35% των Ευρωπαίων πολιτών δεν ξέρουν καν την ενιαία αγορά. Δεν καταλαβαίνουν το νομοθετικό πλαίσιο, τους κανονισμούς μας. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι λιγότεροι κανονισμοί για ε, να μπορέσει το επιχειρηματικό πνεύμα των ευρωπαϊκών λαών να ανθίσει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ντέβα. Τα αγγλικά μου δεν είναι τέλεια. Α, μαθαίνω. λόγο έχει ο κύριος Ντεάντζελης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ενιαία αγορά αποτελεί μεγάλο επίτευγμα και πολύ σημαντικό έτσι ώστε να φτάσουμε στους φιλόδοξους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020. 20 χρόνια ενιαίας αγοράς είναι αρκετά, αλλά έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Γι' αυτό αυτό που έχει σημασία είναι να φτάσουμε σε αυτά που δεν έχουμε επιτύχει. Γι' αυτό θα πρέπει και να κινηθούμε στον τομέα της ενέργειας για να έχουμε μια καθαρή και ασφαλή ενέργεια και πηγές ενέργειας. Να αρθούν τα προσκόμματα, κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία σε αυτή την οικονομική και κοινωνική κρίση που έπληξε την Ευρώπη, διότι έτσι θα φτάσουμε στην καινοτομία, στην ανάπτυξη, στην αύξηση ανταγωνιστικότητας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ντεάντζελης. Η κυρία Μακοβέη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τη Συμφωνία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ενιαία αγορά δημιουργήθηκε για να αυξηθεί η ροή του διακρατικού εμπορίου μεταξύ κρατών μελών χωρίς εμπόδια. Όμως αυτό δυστυχώς δεν συμβαίνει σήμερα. Πρέπει να φροντίσουμε να είναι βέβαιοι οι πολίτες μας ότι υποφελούνται από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι όλοι ανήκουν στην ίδια κοινότητα. Για να πραγματοποιηθεί αυτό θα πρέπει να εμβαθύνουμε έτσι περαιτέρω την ενιαία αγορά. Αυτό θα αυξήσει τον ανταγωνισμό, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Όπως επίσης και τα κοινωνικά ωφέλη, τα οποία χρειάζονται χρήματα. Πρέπει αυτό να το πετύχουμε. Πώς θα το πετύχουμε. Να προωθήσουμε την εναρμόνιση. Να δημιουργήσουμε ας πούμε ένα σύστημα σειροδρόμων, να φροντίσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις λιγότερους κανονισμούς αλλά πιο σαφείς. Η εναρμόνιση είναι ζωτική σημασίας για την ενιαία αγορά αλλά και για τους πολίτες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει ε, ο Άνταμ Βιέλλαν. Στόχος της ενιαίας αγοράς είναι η ελεύθερη διακίνηση των αγαθών, ανθρώπων και κεφαλαίων μεταξύ κρατών μελών, πράγμα που υποτίθεται θα οδηγήσει σε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Όμω, οι έχουν προ... οι πολίτε έχουν πρόβλημα με την λειτουργία αυτή τη αγορά, κυρίω λόγω κάποιων κενών νομικών και ενημέρωση. Υπάρχει λοιπόν πράγματι ανάγκη να υποβληθεί στην Επιτροπή και στα κράτη-μέλη να υποβληθούν κάποιε συστάσει που θα οδηγήσουν στην ε, εναρμόνιση τη ε, ενιαία αγορά. Γιατί όσον αφορά τα κράτη-μέλη πρέπει να αναγνωριστεί η εναρμόνιση των προσόντων, των ε, ιατρικών υπηρεσιών και των τραπεζικών υπηρεσιών. Θα πρέπει να φτιάξουμε μια λειτουργική ενιαία ψηφιακή αγορά που θα ωφελήσει επιχειρηματίες και καταναλωτές. Ε, στηρίζω την έκκληση να εξυγχρονιστεί η εθνική δημόσια διοίκηση ώστε να εισεχθούν περισσότερες ηλεκτρονικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Επίσης, τη στενή συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου, ε, Συμβουλίου και κρατών μελών για να αυξηθεί η πρόσβαση των πολιτών στην διαδικασία λήψη αποφάσεων. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη χαρά υποστήριξα την έκθεση αυτή και όσο νωρίτερα καταφέρουμε να βελτιώσουμε την ε, ενιαία αγορά, τα πράγματα θα βελτιωθούν για όλους μας για, στον τομέα της ύφεσης, αλλά θα υπάρξει και ανάπτυξη για το μέλλον. Αυτό νομίζω ότι αφορά τις ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών και των επιχειρήσεων, κυρίως των επιχειρήσεων, αλλά οι περισσότεροι πολίτες δεν γνωρίζουν τι είναι η ενιαία αγορά και τι σημαίνει. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει. Παρά τα αυτά είναι πολύ λογικές οι προτάσεις και σαφώς πρέπει να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατόν. Δύο πράγματα θέλω να επισημάνω. Τη χρήση του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Πάρα πολλές επιχειρήσεις δεν εμπορεύονται εκτός του ειδικού τους κράτους, να μην μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον, την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Η Έλενα Μπασέσκου. Ευχαριστώ και εγώ υπερψήφισα αυτή την έκθεση για την ενοποίηση, περαιτέρω ενοποίηση της ενίας αγοράς που έχει μεγάλη σημασία για την ε, ανάκαμψη και την ανάκαμψη καθώς και για την εργασία. Βοηθά ε, στην ελεύθερη κυκλοφορία, γι' αυτό θα πρέπει να απομακρυνθούν όλο ένα και περισσότερα προσκόμματα έτσι ώστε οι πολίτες να μην έχουν προσκόμματα όπως ισχύει στην περίπτωση των Ουρμάνων και που πρέπει να αρθούν. Στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης θα πρέπει να άρουμε τα χάσματα έτσι ώστε να προωθήσουμε την ε, ανάπτυξη, την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την περαιτέρω ενοποίηση της ενιαίας αγοράς. Θα πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος διακυβέρνησης μέσα στα πλαίσια της ε, βελτίωσης της συνεργασίας. Επίσης, αυτό που ε, είναι πρωτεύον για μας είναι η ευημερία, η οικονομική και η κοινωνική των πολιτών. Ευχαριστούμε κύριε Μπασέσκου. Περνάμε τώρα στις ε, διαπραγματεύσεις ε, της εμπορικές με την Ιαπωνία. Τι είναι το λόγο στον κύριο Ντίβα ξανά. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έκθεση. Η Ιαπωνία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος μας μετά την Κίνα. Και η Ιαπωνία είχε επενδύσει πάρα πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παραγωγή οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μου, στο Ρωμανό Βασίλειο, είναι αρκετά μεγάλη. 140.000 θέσεις εργασίας υπάρχουν και αυξάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των Ιαπωνέζικων επενδύσεων. Παρομοίως και εμείς θα πρέπει να επενδύουμε στην Ιαπωνική οικονομία και αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να ζητήσουμε από τους Ιάπωνες να μην ε, επιβάλλουν ποσοτικούς περιορισμούς και δασμούς και να ανοίξουν το δίκτυο διανομής τους στις εξαγωγές μας και τις υπηρεσίες μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ορισμένες φορές να κάνει κανείς διανομή εντός της Ιαπωνίας ε, και πρέπει να αντιληφθούν πως πρέπει και εμείς να έχουμε ίσους όρους ανταγωνισμού για να έχουμε πρόσβαση στην Ιαπωνική αγορά όπως και εμείς τους επιτρέψαμε να έχουν πρόσβαση στην δική μας αγορά και να πουλάνε τα προϊόντα τους. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έκθεση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Δίβα. Ο κύριος Μπίλεν. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία μαζί είναι πάνω από το 1 πέμπτο του παγκοσμίου εμπορίου. Πολλά ποιοτικά ε, οι ιαπωνικά προϊόντα αγοράζονται από τους Ευρωπαίους. Μία συμφωνία, αμοιβαία συμφωνία ελευθερμπορίου θα διευκολύνει τους επιχειρηματίε μας να ε, κάνουν εξαγωγές στην Ιαπωνία. Και η πλειοψηφία των επιχειρηματιών είναι υπέρ των διαπραγματεύσεων. Ζητήματα όπως οι δασμοί, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ανταγωνιστικότητα, και η μη δασμολογικοί φραγμοί θα πρέπει να συστηματοποιηθούν. Ταυτόχρονα βεβαίως πρέπει να δούμε την ε, ανάγκη προόδου και της ε, κατάργησης των μη δασμολογικών φραγμών κάτι το οποίο θα επηρεάσει τη μελλοντική θέση του Κοινοβουλίου. Επίσης, για να μην υπάρξει αχαλήνωτη αύξηση των εισαγωγών, πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, τα διμερεί προστατευτικά μέτρα για το μίσο όπως η αυτοκίνητο βιομηχανία. Εγώ λοιπόν είμαι υπέρ της, ε, του ψηφίσματος. Σας ευχαριστώ, ο κύριος Σόγκορ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχοντας υπόψη την ε, παγκόσμια οικονομική κρίση δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι ε, αποφασιστική παγκοσμίου εμπορίου. Κάποιοι θα πούν πως ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της Ασίας χωρίς να αναφέρουμε καν την Κίνα. Οι χώρες του Ασιαν, Σιγκαπούρη, Μαλαισία, Βιετνάμ, Ινδονησία θα τα πάνε πάρα πολύ καλά σε οικονομικούς όρους. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να αναπτύσσει τις συμπορικές της σχέσεις με αυτή την περιοχή του κόσμου και ειδικά με τις χώρες εκείνες οι οποίες έχουν ε, οικονομίες της αγοράς. Και ένα τέτοιο βήμα θα ήταν μια συμφωνία ελευθερία εμπορίου με την Ιαπωνία. Έχουμε μια ανάλογη συμφωνία με την Νότια Κορία και με βάση αυτή την εμπειρία γνωρίζουμε πως Υπάρχει μεγάλο δυναμικό για αύξηση του εμπορίου και προ τι δύο πλευρέ. Μία κατάσταση αμοιβαία υποφελή. Γνωρίζουμε βεβαίω πω υπάρχουν κάποια εμπόδια όπω οι φόροι, οι δασμοί κτλ. Αλλά αυτό δεν είναι ό,τι πιο δύσκολο να επιληθεί. Νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσουν οι μη δασμολογικοί φραγμοί, αν είναι να έχουμε πραγματικά ελεύθερο εμπόριο. Άρα η Ευρώπη πρέπει να δώσει μεγαλύτερο βάρος εδώ πέρα, ειδικά για τις χώρες αυτές στην ΑΠΑ Ανατολή. Νομίζω πως υπάρχει εδώ πέρα πάρα πολύ μεγάλη δυναμικό για εμπόριο. Σας ευχαριστώ. Κύριος Τάνοκ. Θέλω να σα ε, συγχαρώ για τα εξαιρετικά αγγλικά σα, κύριε Πρόεδρε, να συνεχίσετε. Κάποια μέρα θα προσπαθήσω και εγώ να μιλήσω με στη γλώσσα του Δάντη, αλλά όχι ακόμα. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία να είναι υπερήφανε για αυτή τη συμφωνία που ενισχύει αυτή τη συμφωνία. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο η οικονομία, μια φιλελεύθερη δημοκρατία, έχει υψηλά επίπεδα κατανάλωση. και όπω είπα στου είπαν και οι συνάδελφοι έχουμε μεγάλο εμπόριο με την Ιαπωνία. Πέρσι ε, δισεκατομμύρια ευρώ. Η ελεύθερη διακίνηση αγαθών είναι ο χρονιάς λίθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επωφελούνται και οι καταναλωτές αλλά και οι κατασκευαστές. Πρέπει λοιπόν να επιδιώκουμε τέτοιου είδου συμφωνίες ε, όπου και να τις βρίσκουμε αλλά κυρίως με δημοκρατίες όπως η Ινδία και η Ιαπωνία που μας επιτρέπουν να ενεργοποιήσουμε την οικονομική ανάπτυξη η οποία αυτή τη στιγμή λείπει από την Ήπειρό μας. Τα τελευταία 21 χρόνια από την πρώτη κοινή δήλωση Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση Ιαπωνίας για το εμπόριο και άλλα θέματα, είναι σαφές ότι οι πολιτικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας έχουν συνεχώς ενισχυθεί. Αυτή η συμφωνία, η FTA, μπορεί να θα, ωφελήσει και τι δύο πλευρέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ. Και τώρα δίνω το λόγο στον Άνω Τάκολα. Äänestin myös Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα την συμφωνία αυτή. Είμαστε ούτως ή άλλως ε, ο καθένας ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του άλλου, 150 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι εμπορικές ροές, η Ιαπωνία είναι παρούσα στην Ευρώπη, το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά επίσης σημαντικό είναι και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να είναι παρούσες ε, στην Ιαπωνία. Το σημαντικό λοιπόν είναι η αμοιβαιότητα. Πότε πρέπει να καταργηθούν αυτή τη στιγμή οι δασμοί και η Ευρώπη χρειάζεται ανάπτυξη και πρέπει να βγάλουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα. Επίσης πρέπει να σκεφτόμαστε πως είμαστε μία κοινότητα αξιών. Οι πολιτισμοί είναι διαφορετικοί, αλλά έχουμε ευρωπαϊκές νομίζω αξίες και κάποια πράγματα τα οποία είναι κοινά. Κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα, όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο. Σας ευχαριστώ. Τελευταία εξήγηση ψήφου είναι του κυρίου Κέλλη. Σας ευχαριστώ και πάλι. Πρέπει να πω πως σέβομαι ιδιαίτερα την Ιαπωνία, είναι ένα θαυμάσιο έθνος, πολύ έξυπνη φιλή και δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά και έχουν κάνει πάρα πολύ, σημειώσει πάρα πολύ πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Βέβαια τώρα περνάνε δυσκολίες λόγω του τσουνάμι, της Φουκουσίμα και των λοιπόν γεγονότων αλλά θα τα καταφέρουν και θα προοδεύσουν και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τους βοηθήσουμε. Και αυτό μπορεί να γίνει με τη Συμφωνία ελευθερία. και μια σημαντική πτυχή είναι οι δημόσιες προμήθειες. Θα πρέπει να αλλάξουν τη στάση τους όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες και από πιο, είναι από τα πιο σημαντικά σημεία αυτό για την ε, ελεύθερη αγορά μεταξύ μας. Σημαντικό και για μας και για την Ιαπωνία. Σας ευχαριστώ. Η τελευταία τελευταία τελευταία επεξήγηση ψήφου είναι η κυρία Ζαμπόρσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ζήτησα το λόγο. επειδή ήθελα να αντιδράσω και να πάρω το λόγο σε σχέση με κάποια έκθεση. Ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που υπόθηκαν όταν συζητήσαμε την έκθεση της κυρίας Σνίπερ. Ε, θέλω να πω κάτι σε σχέση με, αυτό, με αυτή την προφορική τροπολογία που θέλησε να υποβληθεί. Ο κύριος Κάσμαν χρησιμοποίησε το δικαίωμα του να πάρει το λόγο για να μας υποτιμήσει. Και πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητά πολύ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλοι έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν σύμφωνα με τη συνείδησή τους λυπάμαι πάρα πολύ για το επεισόδιο αυτό. Ναι, η συνεδρίαση λύεται μέχρι τις 3 το απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας όρεξη.